όσα μας είπατε και την υπόδειξη αυτή. Τα πρακτικά και τα ε, κείμενα που εγκρίθηκαν στις 24 Οκτωβρίου διατίθενται. Έχετε στάσεις, αντιρρήσεις, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά. Ερχόμαστε στις ανακοινώσεις. Αρμόδιες αρχές της ε, Ομοσπονδιακής